Item number 16. Είμαστε στο It is now a pleasure to welcome... Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε εδώ τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Κροατίας, τον κύριο Γκόρνταν Κλίτς Ράντμαν. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή αυτή εξωτερικών υποθέσεων. Την ε, προηγούμενη Τρίτη είχαμε στην Ολομέλεια την παρουσίαση του φιλόδοξου προγράμματος της Κροατικής Προεδρίας από τον Πρωθυπουργό Πλέκοβιτ. Σήμερα έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Ράτμαν, ο οποίος πήγε και στην Επιτροπή σήμερα το πρωί, εμπορίου. Τώρα είναι μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας τις ε, προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής της Προεδρίας σας, που φέρει τον τίτλο «Η Ευρώπη που επηρεάζει τα πράγματα». Θέλω λοιπόν να σας δώσω το λόγο και στη συνέχεια θα έχουμε και 45 λεπτά για να ανταλλάξουμε απόψεις με τους συναδέρφους, να σας ρωτήσουν κτλ. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι και καλωσορίζω και, την, και τους συνεργάτες σας, τους οποίους ε, συνάντησα ήδη σήμερα το μεσημέρι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Μακάλιστερ και είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να είμαι σήμερα μαζί σα, Αλλά τώρα που μίλησα και γερμανικά θα περάσω και στα κροατικά μετά τα αγγλικά γιατί είναι ωραίο να είναι κανεί μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορεί να μιλήσει την ε, επίσημη, μια από τι επίσημες γλώσσες τη. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σα και θα σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά επίσης θα ξεκινήσω και διάλογο μαζί σας για διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα σας φέρνω τους χαιρετισμού του Πρωθυπουργού μας, του κύριου Πλέγκοβιτς. Ήταν μέλος αυτής εδώ της Επιτροπής παλιότερα και για δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε την ε, δύναμη να επηρεάζει τα πράγματα και ε, να ενισχύει τις, ε, τη δράση της σε κλάδους όπως είναι η εξωτερική πολιτική, η πολιτική ασφάλεια, εμπόριο κτλ. Εμείς πιστεύουμε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάζει τα πράγματα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας, ε, εμπορίου, ανάπτυξης, αλλά και μέσω της ανθρωπιστικής της δράσης. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αναρμονίσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Συγχρόνως πρέπει να καταλάβουμε όσο γίνεται καλύτερα τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρο γύρω μας, αλλά και συνολικά στον κόσμο. Μόνο έτσι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσει ως ένας ισχυρός παγκόσμιος παίκτη και κάποιος που φροντίζει για την ασφάλεια, ενισχύει την πολυμερή διάσταση και την διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Η κροατική Προεδρία λοιπόν τονίζει ότι μας ενδιαφέρει καταρχήν να φροντίζουμε για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ε, περιοχή μας, στον περίγυρό μας. Γι' αυτό λοιπόν και θα ε, στοχεύσουμε στη σταθερότητα, την ασφάλεια, την αντοχή και τις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις. Θα προσπαθήσουμε επίσης ό,τι καλύτερο για την διεύρυνση, γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί μια επένδυση για την ε, σταθερότητα και την ασφάλεια αλλά και την ευημερία στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος με χώρες στην επικράτειά της που δεν αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή. Η ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στα, στα Δυτικά Βαλκάνια αντικατοπτρίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα και την ευημερία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Η Κροατία λοιπόν αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά τις προκλήσεις όσον αφορά τη διαδικασία προσχώρησης αλλά και τα ωφέλη από το να είναι κανείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και η Κροατία αποφάσισε ότι η διεύρυνση αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας μας και θα έχουμε και τη διάσκεψη κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου αυτό θα τονιστεί ακόμα περισσότερο. Η αξιοπιστία της Ευρώπης ε, δοκιμάζεται ακριβώς ανάλογα με τις επιτυχίες της να επηρεάσει τον περίγυρό της. πώς θα επηρεάσουμε ευρύτερα, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον περιγυρό μας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ καλούς λόγους να συνεχίσει να δεσμεύεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο για την παγίωσή της και να μην επιτρέψει οι ευρωπαϊκές περιφέρειες να αλλάζουν δρόμο. Συγχρόνω, τα Δυτικά Βαλκάνια από τη δικιά του την πλευρά πρέπει να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσει. Ε, η έναρξη διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με στρατηγικό τρόπο τους πιο κοντινούς της γείτονες. Επίσης θέλουμε να κάνουμε προσπάθειες να βοηθήσουμε τη Βοσνία Ζεγοβίνη στο δρόμο προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μοναδική περίπτωση χώρα, όπου η ευημερία της και η σταθερότητά τη εξαρτάται από τρει διαφορετικού λαούς. Έτσι λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε τα ατομικά δικαιώματα όλων των πολιτών στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Επιπλέον, χρειάζεται περισσότερος δυναμισμός στις διαπραγματεύσεις για προσχώρηση με το Μαυροβούνι και την Σερβία. Και επίσης στο Κωσυφοπαίδιο υπάρχει επίσης μια προοπτική και ελπίδα. Τώρα η Τουρκία είναι μια υποψήφια χώρα και στρατηγικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχέσει μα με την Τουρκία είναι περίπλοκε. Έχουμε τι ανησυχίε μα, αλλά επίση έχουμε και συμφέροντα συγκεκριμένα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη μετανάστευση. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για διάλογο, ρεαλιστικό όμως, με την Τουρκία. Αλλιώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να χάνει βάρος όσον αφορά τις σχέσεις με αυτή τη χώρα που είναι σημαντικός παίκτη στην περιοχή. Ανατολικά η Κροατία σκοπεύει την ε, εταιρική σχέση με τις χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά μας να την ενισχύσει. Ε, στόχος μας είναι να καθορίσουμε τις προτεραιότητες μετά το 2020 και στόχους για την πολιτική μας αυτή. Θα υπάρξει σχετική διάσκεψη τον Ιούνιο εδώ στις Βρυξέλλες και θα είναι εφοσιωμένη ακριβώς αυτό. Θα υπογραμμίσουμε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Οι προσπάθειές μας τώρα προκειμένου να πετύχουμε μια συνολική λύση στην κρίση στην Ουκρανία πρέπει να συνεχιστούν. Παρά τις προκλήσεις, Χρειάζεται διάλογος με την Ρωσία ε, για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ανησυχίας. Το σημερινό πλαίσιο βασίζεται σε πέντε κατευθυντήριες αρχές και σε μία διτή προσέγγιση και συνεχίζει να προσφέρει δυνατότητες για δέσμευση επιλεκτικά. Ε, νοτίως, ως χώρα της Μεσογείου δίνουμε μεγάλη σημασία στην ε, πολιτική μας απέναντι στις χώρες που βρίσκονται νοτίως μας και τις χώρες με τις οποίες συνορεύουμε. Το Ιράκ και το Ιεράν βρίσκονται σε αστάθεια, κάτι το οποίο μας ε, επηρεάζει συνεχώς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνδυάσουμε τις ε, προσπαθειές μας. Και ελπίζουμε ότι η διάσκεψη του Βερολίνου της Κυριακής να αποτέλεσε μια κρίσιμη καμπή Χρειάζονται συνδυασμένες ε, προσπάθειες από όλες τις πλευρές, ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση και επίλυση κρίσεων, όπως επίσης να αντιμετωπιστούν και διάφορες προκλήσεις αναμένουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε σημασία στα θέματα της Συρίας, της Λιβύης, της Ιεμένης, του Ιράκ και του Ιράν και των περιοχών του κόλπου γενικότερα. Ο κόσμος σε αυτές τις περιοχές αξίζει να ζει σε ειρήνη, με σταθερότητα, κάτι το οποίο βέβαια θα ευνοήσει και τη δικιά μας σταθερότητα και ασφάλεια. Η στήριξή μας σε ειρηνικές λύσεις με τη συμμετοχή όλων και βιώσιμες με ανθρωπιστική βοήθεια και σταθερότητα αλλά και ανοικοδόμηση. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, της αντιτρομοκρατίας, της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης και του βιοεξτρεμισμού. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για σταθερότητα και ειρήνη, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και τους πρόσφυγες να επιστρέψουν. Τώρα, οι στόχοι των ΗΕ 2030 και ενισχυμένε προσπάθειες των χωρών μελών για να υπάρχει διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη θα είναι πράγματα που θα έχουμε στους δικούς μας ε, στόχους. Όπως επίσης και συνδυτοποίηση για το οικουμενικό πρόβλημα που είναι η κλιματική αλλαγή. Επίσης, χρειαζόμαστε μια συνολική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωσης για και μαζί με την Αφρική. Και αυτό αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι αναγκαίο προκειμένου η Ευρώπη να μπορεί να επηρεάζει τα πράγματα στον κόσμο. Χρειάζεται μια συνολική στρατηγική, λοιπόν, ε, από και για την Αφρική. Το μέλλον της Αφρικής θα επηρεάσει το μέλλον του κόσμου ολόκληρου χρειαζόμαστε μια εταιρική σχέση μακράς διαρκείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρική που να βασίζεται σε αμοιβαία ενδιαφέροντα. Πολλά επίση μπορούμε να κάνουμε και για τι διατλαντικές μας σχέσεις. Η διατλαντική εταιρική σχέση αποτελεί πυλώνα για την ειρήνη και τη σταθερότητα παγκοσμίω και αποτέλεσε ένα ουσιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής ασφάλειας και ευημερίας. Ανεξάρτητα από τις διαφορές που μπορεί να έχουμε για μερικά ζητήματα, πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπέρ της σταθερότητας στην γειτονιά μας και να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ μας απειλές και προκλήσεις όπως είναι η τρομοκρατία, η μη διάδοση όπλων, η μετανάστευση και η ενεργειακή ασφάλεια. Στην Ασία τώρα επικεντρωνόμαστε στην διασυνδεσιμότητα και θέλουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Κίνα. Η συνδεσιμότητα είναι ο δεύτερος πυλώνας των προτεραιοτήτων ε, της Προεδρίας ε, σε όλες τις πτυχές της, την οικονομική, υποδομών, ψηφιακή και ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους τους ίδιους. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο εργαλείο για συνεργασία σε έναν κόσμο που είναι όλο και πιο κατακαιρματισμένος. Δύο διασκέψεις κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας θα λάβουν χώρα φέτος, 17 συν 1. Και πρέπει να υπάρξει ενότητα, συνοχή και αποτελέσματα και για τις δύο πλευράς. Η Προεδρία μας θα συνεχίσει να ενισχύει τη στρατηγική μας εταιρική σχέση επίσης και με τη Λατινική Αμερική. Η Ήπειρος αυτή αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και αστάθεια, τόσο πολιτική όσο και οικονομική, που δυστυχώς ενισχύεται με τον καιρό. Εμείς εδώ θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην Βενεζουέλα και θέλουμε να βοηθήσουμε τις γείτονες χώρες να αντιμετωπίσουν τις μεταναστευτικές πιέσεις. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ και σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι η συνεργασία μας με σημαντικούς εταίρους. Καναδάς, Μεξικό, Βραζιλία, Ινδία, Νότια Αφρική, Κορέα, Ιαπωνία και Αυστραλία. Ζούμε σε ένα κόσμο που αλληλοεξαρτάται όλο και περισσότερο. Γι' αυτό οι σχέσεις αυτές έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά τώρα την ασφάλεια και την άμυνα. Και εδώ θέλουμε να πετύχουμε περισσότερη συνοχή ε, στο τομέα των πρωτοβουλειών και των μηχανισμών μας. Θα ενισχύσουμε ακόμα τη συνεργασία μας με τον ΝΑΤΟ και θα πιέσουμε για να έχουμε την δικιά μας άμυνα ενισχύοντας την έρευνα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Να μην ξεχνάμε και τη μη πτυχή της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης μας προσέγγιση. Εν κατακλείδη, η κρατική προεδρία έρχεται σε στιγμές ε, δύσκολες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Κροατία. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πριν από μερικά χρόνια ότι η Κροατία θα ήταν ανεξάρτητη χώρα και τώρα έχουμε ήδη τόσα χρόνια μετά την αναγνώριση της σύγχρονης Κροατίας δεν είμαστε μόνο ε, μέλος στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προεδρεύουμε και όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ίσως να το... να μην το βλέπετε, αλλά πραγματικά είμαστε περήφανοι. Γιατί για την Κροατία είναι μια ιστορική στιγμή να βρίσκεται επικεφαλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει αναλάβει την Προεδρία της. Αποτελεί προνόμιο για μας. Η Κροατία ολοκλήρωσε όλους τους στόχους για την εξωτερική πολιτική. Τώρα στην Προεδρία μας οι προτεραιότητές μας δεν είναι μόνο προτεραιότητες της Κροατίας, είναι ευρωπαϊκές προτεραιότητες, είναι οι δικές σας προτεραιότητες. Γιατί εμείς τις δικές μας τις καλύψαμε. Φυσικά υπάρχουν κάποιες ακόμα, όπως συμμετοχή στο Σέγγεν, στην Ευρωζώνη, γιατί η Κροατία μπορεί κάλλιστα να είναι μέλος και σε αυτά τα όργανα. Εξού και έχουμε ακόμα περισσότερα κίνητρα και νιώθουμε ακόμα πιο φιλόδοξοι για να εκφράζουμε και να εκπροσωπούμε την Ευρώπη στον κόσμο όσο γίνεται καλύτερο. Ο κόσμος είναι γεμάτος προκλήσεις. Γι' αυτό και η Ευρώπη πρέπει να είναι ισχυρή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια λαλάπο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή σας. Έχουμε ακόμα περίπου 35-40 λεπτά στη διάθεσή μας για μια ανταλλαγή απόψεων. Προτείνω να έχουμε ένα πρώτο γύρο παρεμβάσεων από τις πολιτικές ομάδες και μετά και ένα δεύτερο, αν συμφωνείτε. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το ΕΛΚ κυρία Σόφκο ή κύριος Γκάλαρ. Ποιος θέλει να πάρει πρώτο το λόγο. Γέλανα Σόφκο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάλαρ που μου επιτρέπει να μιλήσω πρώτη. Θα μιλήσω στα κρατικά, εφόσον έχουμε μια τέτοια τιμή να έχουμε την Προεδρία και για πρώτη φορά έχουμε εδώ μαζί μας έναν ε, Κροάτι Υπουργό Εξωτερικών. που συντονίζει την ε, εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργέ, καλώς ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. σε ένα χώρο νέων ιδεών σε ό,τι αφορά το συντονισμό των, της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων όσα μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στους επόμενους έξι μήνες για να πετύχει τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ειρήνη. Στη Σύνοδο Κορυφής που θα λάβει χώρα στην Κροατία κατά τη διάρκεια της Κροατικής Προεδρίας, Σε αυτή τη Σύνοδο λοιπόν, θα δούμε τη συζήτηση για το καθεστώς της Βορείου Μακεδονίας και της Αλβανίας μετά το γαλλικό non-paper. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα στο οποίο καταδικάζει την μη έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Θεωρούμε ότι ε, θα μπορέσετε εσείς ε, να διευκολύνετε τα, πράγματα προκειμένου να υπάρξει θετικό μήνυμα από τη Σύνοδο Κορυφής ε, και να ξεμπλοκάρει αυτό το ζήτημα στο Συμβούλιο. Προκειμένου αυτές οι δύο χώρες να μπουν στις διαπραγματεύσεις εν ώψη περαιτέρω διεύρυνσης. Πιο συγκεκριμένα όμως θα ήθελα να ρωτήσω τι θα κάνετε με τη Βοσνία Ρεζεγοβίνη που παραμένει η πιο ευάλωτη χώρα από τις έξι των Δυτικών Βαλκανίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλιστα, έχει υιοθετήσει τέσσερα ψηφίσματα για τη Βοσνία-Ριζεγοβίνη. Τα οποία, μάλιστα, ψηφίστηκαν με μεγάλη διαφορά. Γνωρίζω ότι τα ψηφίσματα βεβαίως δεν είναι δεσμευτικά, αλλά τι νόημα έχει να υιοθετούμε τέτοια ψηφίσματα εάν ε, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη δεν ε, θέλουν να λάβουν υπόψη τις θέσεις μας. Κάποιες από αυτές τις συστάσεις ε, σίγουρα θα συμπεριληφθούν στη συζήτηση κατά τη διάρκεια της ε, συζήτηση Υποκρατική Προεδρία, Ιδίω ό,τι αφορά το συνταγματικό σκέλο που έχει να κάνει με την Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τον Ίνο Πίτσουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας. Χαιρετίζουμε τις ε, προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Κροατία είναι το νεότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον έχει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δίνει το καλό παράδειγμα και στους υπολείπους. Όμως υπήρξαν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διεύρυνση, με βέτο για τι διαπραγματεύσει, σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία πέρσι. Το Κοινοβούλιο ανταπάντησε με ένα ψήφισμα ε, όπου καταδίκασε αυτή την απόφαση και ξέφρασε τη στήριξη προς τη διαδικασία διεύρυνσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανακοίνωσε μια νέα μεθοδολογία στις αρχές του επόμενου μήνα Εσείς ε, ως προεδρεύουσα χώρα, τι προτίθεστε να κάνετε εν ώψη τη ε, Συνόδου Κορυφής στο Ζάγκρεπ για να πετύχουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων με αυτές τις δύο χώρες. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορεί να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία με μια πιθανή συνεργασία μέσω των συστάσεών μας προς το Συμβούλιο, τις οποίες μάλιστα συνέταξα. Την Κυριακή οι ηγέτε ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν επί μια εκεχηρία ε, στο Βερολίνο για τη Λιβύη. Όμω η ειρήνη ακόμα είναι ιδιαίτερα ε, ασταθή και πολλέ προσπάθειε πρέπει να υπάρξουν ακόμα για τη διασφάλιση τη ειρήνη. Καθότι προέρχομαι από τη Μεσόγειο και ξέρω πόσο σημαντική είναι η ειρήνη σε αυτή την περιοχή, πώ μπορούμε εμεί να προάγουμε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ω διαμεσολαβητή σε αυτέ τι συζητήσει. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας, όσο γίνεται λιγότερες κρίσεις και όσο γίνεται περισσότερες λύσεις στα προβλήματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πίτσουλα. Ο κύριος Κιουτσούκ από το Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ. Φέτος ξεκινήσαμε πολύ δυνατά σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική αλλά και η Κροατία ως προεδρεύουσα χώρα. Μ' ακούτε? Εάν ακολουθήσουμε λοιπόν τα όσα είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν, είχε θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους για τα Δυτικά Βαλκάνια, πολύ καλά όλα αυτά, χαιρόμαστε. Όμως, έχει έρθει η ώρα να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν, ακόμα και από την περσινή χρονιά. Δεν πρέπει να κάνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ε, προσιλωμένη στην ε, διεύρυνση και στην ε, ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες υποσχέσεις. Είναι σημαντικό να θέτουμε προτεραιότητες, το ξέρω και από την Βουλγαρική, Βουλγαρική Προεδρία. Τότε και πάλι είχαμε τα Δυτικά Βαλκάνια ως προτεραιότητα. Αλλά και στι προτεραιότητε που θέτουμε πρέπει να υπάρχει επίπεδο φιλοδοξίας. Υπάρχουν προ... διάφορες προτάσεις επί τη μεθοδολογία. Μία προτείνει η Γαλλία, Ε, μία προτείνει η Γαλλία, μια άλλη ομάδα χωρών προτείνει μια άλλη. Δεν ξέρω, ίσως υπάρχει και μια κρατική μεθοδολογία που θα θέλετε να, να προτείνετε. Να έχετε μια δική σας προσέγγιση. Μετά, για τη Σύνοδο Κορυφής ε, του Ζάγκρεπ θα είναι πολύ σημαντική. Η εμπειρία μας δείχνει ότι όλες αυτές οι σύνοδοι κορυφής όλο ένα και ευθύνουν ε, σε σημασία. Αν θυμάστε το 2003 στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ σημαντική, μετά όμως ε, στην ε, Σόφια είχε λιγότερη σημασία πια. Δεν υπήρξε δικός χάρτης για παράδειγμα, για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι λοιπόν ο στόχο της ε, Κροατικής Προεδρίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ζάγκρεπ. Και τρίτον, σωστά είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι. Θα υπάρξουν ε, συναντήσεις ε, υπό, τις, υπό Κροατική Προεδρία. Υπό Βουλγαρική Προεδρία είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση στην πόλη Βάρνα με πολύ σημαντικά ζητήματα που συμφωνήθηκαν εκεί. Αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κιουτσούκ. Ο κύριος Μπουτικόφερ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Με χαρά άκουσα να τονίζετε το ρόλο της ε, σωστής διασύνδεσης ως πυλώνα της εξωτερική πολιτικής που θα επιδιώξετε να ενισχύσετε στην Προεδρία σα. Ήθελα να μου πείτε πώς αυτό σκοπεύετε να το προωθήσετε όντω και πώς σκοπεύετε να υλοποιήσετε αυτή την προτεραιότητα στο πλαίσιο του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Διότι εάν δεν επενδύσουμε εκεί που έχουμε υποσχεθεί να επενδύσουμε, στην ε, διασύνδεση, και όλα αυτά παραμένουν λόγια, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Έπειτα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Μόλις το ρώτησε ο συνάδελφος από την ομάδα Renew. Τι μεθοδολογία θα ακολουθήσετε. Έχετε σημειώσει τις προτάσεις για αλλαγή μεθοδολογίας που έχει εκδώσει ως σύσταση η ΕΕΔ Είστε έτοιμοι να ανοίξετε ενδεχομένως την πόρτα σε μια από τις δύο χώρες που είχαν κάνει την αίτηση Βόρεια Μακεδονία ή κάθετος και Αλβανία ή επιμένετε καμία από τις δύο χώρες να μην περάσουν σε προενταξιακές διαπραγματεύσεις προς τη στιγμή. Και τρίτον, Σε αρκετέ περιπτώσει αναφέρεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ούτε, μάλλον δεν το αναφέρεται ούτε στα πλαίσια του διαλόγου με την Τουρκία, ούτε στο πλαίσιο τη συζήτηση με την Αφρική, ούτε με την Κίνα. Τι ε, κατεύθυνση θα δώσετε στα ανθρώπινα δικαιώματα ως γνώμονα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για μετά για τους εσωτερικού μας διχασμούς οι εξωτερικοί παραγοντές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εσωτερικές διαστάσεις απόψεων. Λόγου χάρη η Κίνα προσπαθεί να εκφοβήσει μια χώρα σαν τη Σουηδία. Είναι πρόσφατο. Τι θα κάνετε για να ξεπεράσετε τέτοιου είδους διχασμούς και να ενισχύσετε την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Να ενισχυθούν χώρες οι οποίες έχουν βρεθεί απομονωμένες και εκτεθειμένες γιατί δέχονται επιθέσεις από εξωτερικούς παράγοντες. Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο πρώτος γύρος. Η ID, ε, οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές και η δεν θέλουν το λόγο. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος. Θέλετε να απαντήσετε τώρα και μετά να έχουμε ένα δεύτερο γύρο. Τι προτιμάτε. Θέλετε να απαντήσετε τώρα. Ωραία. Ευχαριστούμε. Κυρία Ζόφκο, η δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανία βρίσκονταν ε, στην ε, πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της κρατικής προεδρίας Τώρα αναφέραμε την ε, έναρξη διαπραγματεύσεων και την έναρξη ακριβώ τέτοιων διαδικασιών. Στην περίπτωση τη Βόρεια Μακεδονία υπήρχε το θέμα τη ονομασία τη χώρα. Αυτό έχει επιληθεί. Ήταν η μόνη βασική προϋπόθεση που έπρεπε να εκπληρωθεί. Το επέλυσαν με την Ελλάδα και νομίζω ότι τους αξίζει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία επίσης έχει επιτελέσει πρόοδο και υποστηρίζουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις δύο αυτέ χώρε. Ως προς τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπως είπα στην αρχική μου εισήγηση, είναι χώρα γειτονική της Κροατίας. Έχουμε κοινή ιστορία και υποστηρίζουμε την Ερζεγοβίνη, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, βάσει των συμφωνίων του Ντέιτον που θέλουμε να λειτουργεί εύρυθμα. Ε, θέλουμε να υπάρχει ένα σύστημα που να εγγυάται την ε, ειρηνική συνύπαρξη των τριών εθνοτήτων που ζουν εκεί. Βοσνίων, Σέρβων και Κροατών. Είναι βεβαίως σημαντικό για μας όλοι οι συμμετέχοντες πληθυσμοί στη Βοσνία Ζεγοβίνη να συμφωνούν προς την πολιτική τους εκπροσώπηση, διότι η πολιτική εκπροσώπηση του καθενός ατομικά είναι ε, προϋπόθεση και θεμέλιο της δημοκρατίας και είναι και συνιστόσα των ευρωπαϊκών προτύπων. Η Κροατία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ισότητα, τα ίσα δικαιώματα, την ισοτιμία των τριών εθνοτήτων που συγκατοικούν στην Βοσνία Ζεγοβίνη. Ως προς, την, ως προς τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου, το λέω εκπροσωπώντας όχι μόνο την Κροατία, ολόκληρο και την Ένωση πιστεύω, Βεβαίω τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική φωνή, πρέπει να την αφουγκραστεί κανείς και έχουμε ενισχύσει και τη θέση μας για τα θέματα αυτά. Έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε γιατί είναι προς όφελος όλων μας να υποστηρίξουμε την ευρωατλαντική πορεία της Βοσνίας Αζεγοβίνης. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Τονίνο Πίτσουλα, ο οποίος ήταν υπουργό Εξωτερικών πριν από 20 χρόνια όταν έγινε η πρώτη συνάντηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στις 24 Νοεμβρίου 2001. Μετά την Σόφια, το Ζάγκρε, πιστεύω ότι θα είναι επόμενη ε, τοποθεσία για ένα τέτοιο ραντεβού και ίσως να καταφέρουμε κάθε χρόνο παραχρόνο να οργανώνουμε μια τέτοια σύνοδο. Όλες οι κροατικές κυβερνήσεις έχουν κάνει πολλά. Η τωρινή όμως με τον Άντρε Πλένκοβιτς έχει κάνει τα περισσότερα. Οπότε τώρα πρέπει εμείς να προεδρεύσουμε στο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι προβλέπετε, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. για τα Δυτικά Βαλκάνια, Μα συγχωρείτε, αλλά υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα ε, με τη διερμηνία από τα αγγλικά. Δεν χρειάζεται διερμηνία γιατί μιλώ βουλγαρικά, λέει ο μιλητής. Με συγχωρείτε. Συνάδελφοι, όπως εξήγησα στον συνάδελφο μου από τη Βουλγαρία στα βουλγαρικά, τον ευχαρίστησα για την ερώτησή του. Ρώτησε για, την, ε, για το όραμα της Κροατίας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και τι θα κάνει η Κροατία προκειμένου να έχουν μια καλύτερη θέση οι χώρες αυτές. Εγώ έλεγα ότι θα πρέπει να διοργανώνονται σύνοδοι, αλλά όχι μόνο για λόγους πανηγυρικούς και για να οργανώσουμε ακόμα μια εκδήλωση, αλλά να οδηγούν σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Αυτό είναι ο στόχος μας και η πρώτη μας προτεραιότητα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρθηκαν αρκετές φορές νομίζω. Αναφέρθηκαν για την Κροατία είναι μείζον ζήτημα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω δικαίου, ισότητα, ίση μεταχείριση. Θέλουμε να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους τους τομείς του τομεί πολιτική και εξωτερική δράση και να δείξουμε την ενότητα τη εξωτερική μα δράση και τη συνοχή τη. Και για την Αφρική, έχω αναφέρει ποιε είναι οι προσδοκίε μου για την Αφρική και τι πέντε χώρε του Σαχέλ που χρειάζονται τη βοήθειά μα. Χρειάζονται βοήθεια. Ε, η κατάσταση πραγματικά μας κάνει να ανησυχούμε. Έχουν ζητήσει όχι μόνο ηλική βοήθεια και οικονομική, αλλά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα σε αυτήν την περιοχή της Αφρικής. Βεβαίως, για το πρόγραμμα δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Αυτό θα πρέπει να την κατοπτρίζει και την αντιμετώπιση των νέων διεθνών προκλήσεων, όπως τις κλιματικές αλλαγές, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεχνητή ευφία, αλλά και τη μετανάστευση, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και γυναικών, αυτά θα πρέπει να ε, λαμβάνουν όλο ένα και μεγαλύτερη θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων μας. Για την Τουρκία. Συμφωνώ. ανέφερα την Τουρκία γιατί ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν εκεί. Ωστόσο, η Τουρκία είναι σημαντικότατος παράγοντας ε, με γεωπολιτική βαρύτητα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και με τη χώρα αυτή. Ε, φυσικά θα πρέπει να κοιτάξουμε να πείσουμε Και μας ανησυχεί η κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Γι' αυτό παρακολουθούμε και καταδικάζουμε τα έκτροπα που μπορεί να συμβαίνουν εκεί. Όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει πώς μπορεί να επηρεάσει τρίτες χώρες όπως την Τουρκία πώς μπορεί εκεί να βοηθήσει στην προστασία και την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αντιπροσωπείες της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι ένας σημαντικός πρωταγωνιστής, αλλά θα πρέπει να δείξουμε την προθεμία και τον ενεργό ρόλο που αναλαμβάνουμε. Αυτή είναι και η δουλειά του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και όλων ημών. Εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λόγου χάρη. Και όλα τα άλλα θεσμικά όργανα πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε σταθερά και να είμαστε δραστήριοι προς αυτό το σκοπό η κυρία Νικολίνα Μπρένιετσκ, η οποία είναι επιτετραμένη υπουργό για τα θέματα αυτά, θα μα εκπροσωπήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα είναι εδώ για να συνομιλήσετε, θα είναι παρούσα και θα κοιτάξει να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όσο αφορά την Κίνα, σημαντική τρίτη χώρα. Πρέπει να δούμε την Κίνα ως ένα σοβαρό και βαρύνοντα ε, πρωταγωνιστή. Θέλουμε από τη μια να τους ασκούμε λοιπόν πίεση για συγκεκριμένα ζητήματα, θέλουμε όμως να μπορούμε και να έχουμε διάλογο μαζί τους Για την Ξέν Γιάνγκ έχουμε την ε, ευθύνη με την αντιπροσωπεία μας εκεί να προωθούμε και τις τρεις πυλώνες ε, του ΟΗΕ, της πολιτικής του ΟΗΕ για την Κίνα, την ε, πολιτική σταθερότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σταθερότητα. Είναι φυσικά προϋπόθεση για τις διμερείς μας σχέσεις ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Νωρίτερα μου είπε κάποιο από τη Σουηδία, μια βουλευτή από τη Σουηδία το ίδιο πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει αλληλεγγύη και προς τη Σουηδία εάν υπάρξουν οποιασδήποτε διαφορές έστω και διμερεί, και να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται στήριξη και αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Υπουργέ. Τώρα να πάμε στο δεύτερο και τελικό γύρο, να δώσω το λόγο σε όλους τους άλλους συναδέλφους που τον ζήτησαν. Στον κατάλογό μου έχω από το ΕΛ τον κύριο Γκάλερ, τον κύριο Πλέντσακ, τον κύριο Μιγιανμόν, τον κύριο Κρίσταν, Φρίντες, Νόιζλ, ε, Γκλουξμαν, ε, Ντέλη. Νομίζω αυτά είναι τα ονόματα. Σε 17 λεπτά θα έρθει ο κύριο Στόλτεμπεργκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Εδώ είμαι, τελείως δεξιά. Εδώ, εδώ. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή και από τη δική μου την πλευρά χαίρομαι που είστε υπερήφανο να έχετε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, κάθε τύχη λοιπόν στο εξαμεινό σα. Ε, είχαμε το πρωί ακρόαση για τα θέματα της Λιβύης και τη σχετική σύνοδο. Υπάρχει ένα συγκρατημένο, μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τα θέματα της Λιβύης και ένα ε, θέμα κρατήσαμε εδώ. Το τι θα γίνει με την εξακολούθηση της επιχείρησης Σοφία Ακούσαμε πολλές δηλώσεις συναδέλφων και θέλαμε και εσείς να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Η επιχείρηση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και είναι κάτι που δεν έχουμε κάνει αρκετά ως τώρα να κοιτάξουμε να ελέγχουμε εάν τηρείται το εμπάργκο των όπλων. στις συγκεκριμένες ε, συγκυρίες και περιστάσεις θα πρέπει να δούμε μήπως χρειάζεται έλεγχος όχι μόνο από ρωσικά σκάφη ή κάποιο σκάφος του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση και μετά, μετά την ε, σύνοδο του Σαββατοκύριακου. Έχετε την εντύπωση ότι μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών κρατών, τέλος πάντων των 27 ενωπομινάντων, υπάρχει μια ομοιογενής θεώρηση του θέματος της Λιβύης. Ο στρατηγός Χαφτάρ υποστηριζόταν από τη Γαλλία και τέλος πάντων εκεί είχε συμπάθειες. Οι Ιταλοί υποστήριζαν τον άλλο στρατηγό. Ε, Πώς θα ε, κινηθούμε λοιπόν σε σχέση με την κυβέρνηση και με ποιες δυνάμεις θα την υποστηρίξουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ Υπουργέ. Θέλω να θίξω το θέμα των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της Κροατίας και Βοσνίας Ζεγοβίνης. Πάντα μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά το κόσμο ε, και πώς θέλουμε να τα προστατεύουμε, αλλά είναι θέμα αξιοπιστίας μας να συμμορφωνόμαστε εμείς ήδη με τα ανθρώπινα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, στις χώρες μας. Και θέλω λοιπόν να θέσω το ζήτημα της συμπεριφοράς μας απέναντι στους πρόσφυγες αυτούς έξω από τα σύνορα της Κροατίας στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Υπήρξε βία και από τις κροατικές αρχές και στα σύνορα με αποδείξεις. Και δεν τα λένε αυτά μόνο μη κυβερνητικέ οργανώσεις στα μέσα ενημέρωσης, αλλά ε, τα είπε και ο τέος πρόεδρος ότι η αστυνομία τα ταπείνωσε πρόσφυγες, δεν είχαν στη διάθεσή τους τίποτα, τους πήραν τα παπούτσια, τα χρήματα, τα πάντα. Η βία και η πίεση με βία πολλές φορές να πάνε πίσω είναι καθημερινότητα. Η Κροατία θέλει να γίνει μέλος της Σέγγεν. Πώς θα γίνει όμως αυτό πώς θα υπάρχει ελεύθερη διακίνηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έχουμε τέτοιες πρακτικές. Εγώ πιστεύω ότι τέτοια προσχώρηση στο Σέγγεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Τι να κάνουμε λοιπόν και τι θα κάνετε για να σταματήσει αυτή η συμπεριφορά, θα ελέγξετε τα σύνορα ώστε να ερευνώνται σωστά οι παραβιάσεις που γίνονται όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στους πρόσφυγες. Ο κ. μισή λεπτό το πολύ γιατί στις και μισή θα πρέπει να σταματήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω και εγώ στη γλώσσα μου. Θα ήθελα μια εξήγηση, μια διευκρίνηση τέλο πάντων. Στο πρώτο τμήμα, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε ε, στις προτερότητές σας και στα πλαίσια των συνταγματικών αλλαγών βάσει των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να ξέρω αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η πολιτική εκπροσώπηση για τις τρεις χώρες στη Βοσνία Ριζεγοβίνη σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί πάλι ε, μια επικράτεια ή ότι η, θα ληφθεί υπόψη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι μία από τις καλύτερες τελευταία. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ότι διασφαλίζουμε πολιτικά δικαιώματα συνολικά, σε συνολικό επίπεδο, ή σημαίνει τρίτη οντότητα. Σαν Dayton 3 και όχι Dayton 1. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκρόσλεϊ. Ελκ Σαν Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Λέει κυρία Κλάβακ. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, οι σχέσεις μας είναι πολύ σημαντικές γιατί θέλουμε την ενίσχυση και την πολιτική προσέγγιση. Έχουμε την Αρμενία, το Ζερβαϊτζάν, την Λευκορωσία, Μολδαβία και και την Ουκρανία. Σήμερα το πρωί εμείς ακούσαμε την παρουσίαση των σχετικών εκθέσεων. Και είναι σαφές ότι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατολικά και στον Κάφκασο είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα, η ευημερία, η ειρήνη και το κράτος δικαίου. Χάρη τώρα στη Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθερότητας μετά το Dayton και τις υπόλοιπες συμφωνίες, η Μολδαβία και η Γεωργία επέρασαν στο επόμενο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, θέλω να ξέρω με ποιο τρόπο η Κροατική Προεδρία ε, σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα της ανατολικής εταιρική σχέσης και πώς θα αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και τις νέες συνθήκες κάτω από τις οποίες ε, ζουν τώρα αυτές οι χώρες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαυρίδης είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εδώ. You might need your headphones. Thank you. Στην εισαγωγή σας είχατε τονίσει ότι τη σημασία για, θα το διαβάσω στα αγγλικά, fighting terrorism, radicalization and extremism. Ας είμαστε όμως συγκεκριμένοι για το τι μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουρκία. Η χώρα βρίσκεται υπό συγκαλυμμένη δικτατορία, υπό τις διαταγές του μονάρχη, του νέου σουλτάνου οι λαοί και ειδικά οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένουν από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεσματικότητα και να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικότητες. Από ό,τι κατάλαβα, ακούγοντα σας και νωρίτερα σε άλλη επιτροπή και τώρα, περίπου προτείνεται τη συνεργασία ή το engagement, αν το κατάλαβα σωστά, το οποίο έχει δοκιμαστεί και έχει αποτύχει με την Τουρκία. Επιπλέον όμως, αυτό έχει δύο μεγάλα λάθη όχι μόνο έχει αποτύχει, ήδη λαμβάνοντας υπόψη την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας και του Ερτογάν στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά σε σχέση με την Κυπριακή ΑΟΣ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο εσείς προεδρεύετε, έχει αποφασίσει συλλογικά και ομόφωνα να προχωρήσει σε άλλη πολιτική, την αποκοπή κονδυλίων και την επιβολή κυρώσεων. Επομένως, αναμένω κύριε Υπουργέ, να μας πείτε πώς θα κινηθείτε σε αυτή την πορεία για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό τον οποίον προάγει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο προτού κλάψουμε επί ερυπείων όπως κλάψαμε στη Συρία, στην Κύπρο, στο Αφρίν, στη Λιβύη και αλλού. Thank you, Mr. Milan Ευχαριστούμε, ο κύριος Μιλανμόν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Χάρηκα που αναφερθήκατε και στις χώρες γειτονία του Νότου και όχι μόνο ανατολικά. Έγινε διάσκεψη για την Λιβύη, αλλά υπάρχουν ε, και άλλες σημαντικές χώρες. Εκεί δεν υπάρχει μόνο η Λιβύη και λιγότερο προβληματικές ίσως, όπως είναι το Μαρόκο, Αλγερία κλπ. Και ελπίζω να δώσετε την ίδια σημασία και σε αυτές τις μεσογειακές χώρες. Χαίρομαι επίσης που τα τελευταία που είπατε είχαν να κάνουν με τη Λατινική Αμερική, γιατί συχνά τις ξεχνούν οι προεδρίες. Η Λατινική Αμερική αποτελεί ένα φυσικό εταίρο και σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάμε ότι η Βενεζουέλα εξακολουθεί να ε, βρίσκεται στην προσοχή μας. Ο κύριος Μπορέλ αύριο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Γκουαϊντό και η Βενεζουέλα θα ήθελα να παραμείνει προτεραιότητα και κατά τη διάρκεια της Κροατικής Προεδρίας για να στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί και για να λυθούν μέτρα, εάν γίνεται ακόμα και κυρώσεις κατά του καθεστώτος του Μαδούρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Νόιζελτ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, εδώ κάθομαι. αναφερθήκατε και παρουσιάσατε ε, πολλές διασκέψεις, συναντήσεις. Δεν άκουσα όμως κάτι. Γιατί συνήθως όταν υπάρχει προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί γίνεται η μικτή συνέλευση με τις χώρες ΑΚΕ. Και θα ήταν ο ρόλος της Κροατίας τώρα να φιλοξενήσει τη διάσκεψη αυτή που συμμετέχουν πάνω από 100 χώρες. Μέχρι τώρα άκουσα ότι η κυβέρνησή σας διστάζει. Οπότε ρωτάω, τι θα γίνει με την ε, JPA, θα την φιλοξενήσει η Κροατία ή όχι. Τέλος, Ντέλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που ήρθατε και μας μεταφέρατε τις σκέψεις σας όσον αφορά την διεύρυνση. Δεν λέω ότι πρέπει να ξανεφεύρουμε τον τροχό, αλλά τι θα γίνει με την Προεδρία σας. Ε, πρώτα θα πρέπει να πείσετε τους πιο σκεπτικιστές και μετά θα πρέπει να ανακτήσετε την εμπιστοσύνη από τα Δυτικά Βαλκάνια. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο η πρώτη πλευρά είδα ότι γίνονται συναντήσεις υψηλού επίπεδου των υπουργών σας με τον Πρωθυπουργό Μακρόν και τα λοιπά. Πόσο φιλόδοξο είσαστε και πόσο αισιόδοξο μάλλον, συγγνώμη, αισιόδοξο είσαστε ότι θα τα καταφέρετε στην διάσκεψη του Μαΐου όσον αφορά ε, την διεύρυνση. Ωραία. Τα δικά σας σχόλια, κύριε Υπουργέ. Θα καθυστερήσει 5 λεπτά ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, οπότε σε 10 λεπτά πρέπει να μα έχετε απαντήσει. Θα τα καταφέρετε, 10 λεπτά. 10, 10, το πολύ 10. Ευχαριστώ πολύ. Γερμανικά. Με την επιχείρηση Σοφία, Ήδη από χθε το συζητήσαμε στο πλαίσιο των εξωτερικών υποθέσεων ότι πρέπει η επιχείρηση Σοφία να συνεχιστεί να ανανεωθεί. και να προχωρήσει η διαδικασία. Και να προχωρήσουμε. Έχουμε ήδη πετύχει αρκετά. Έχουμε ήδη κάποιες προϋποθέσεις για την κατάπαυση πυρός. Πρέπει όμως να εφαρμόζεται σωστά το εμπάργκο των όπλων. Σε κάποιο βαθμό λοιπόν κάτι έχουμε ήδη πετύχει, όμως πρέπει να γίνει περαιτέρω πρόοδος. Χρειάζεται βεβαίως χρόνος και διπλωματικές προσπάθειες και όλα τα σχετικά, αλλά ήδη έχουν όλοι κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια και συνεχίζουν. για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στο θέμα της μετανάστευσης και όσον αφορά την ε, Βοσνία, πρέπει να σας πω ότι η Κροατία προστατεύει τα εθνικά σύνορα που αποτελούν και εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους παράτυπους μετανάστες και τα μεταναστευτικά ρεύματα. Οπότε με περηφάνεια η Κροατία προστατεύει τα σύνορά της από τα φαινόμενα αυτά. Κάτι το οποίο είναι και υποχρέωση κάθε δημοκρατικής χώρας. Οπότε εμείς προστατεύουμε την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης τελικά. Ο Σλοβαίνος συνάδελφος έθεσε επίσης ένα ερώτημα για την αντιπροσωπευτικότητα. Εμείς υποστηρίζουμε το δικαίωμα κάθε πολίτη που ζει μέσα σε ένα δημοκρατικό χώρο το δικαίωμά του να εκλέγει αντιπροσώπους. Εγώ δεν μιλάω εδώ πέρα για μια νέα σύλληψη ή για μια νέα εδαφική επικράτεια. Όχι, η Κροατία ήταν η πρώτη που αναγνώρισε την ανεξαρτησία και την εδαφική ακαιρότητα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η ανατολική εταιρική σχέση βεβαίως και αποτελεί προτεραιότητά μας. Πρόκειται όχι μόνο για την δημιουργία της αντίληψης ότι θέλουμε προσέγγιση, αλλά ότι θέλουμε προσέγγιση με τους ανατολικούς εταίρους μας επίσης, όχι μόνο με τα Δυτικά Βαλκάνια. Εξού και γίνεται και η προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση της δημοκρατίας προκειμένου να παγιωθεί η ικανότητά τους και να μπορέσουν έτσι οι χώρες αυτές να υιοθετήσουν τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου η ευρωπαϊκή τους προοπτική να ενισχυθεί. Και προτείνουμε και περισσότερο άνοιγμα. Έρχομαι τώρα στη Μεσόγειο. Η Κροατία τον Απρίλιο στην πόλη Σίμπενικ που είναι στις Αδριατικές Ακτές θα φιλοξενήσει μία διάσκεψη για τη Μεσόγειο. Εκεί θα συμμετέχουν όλες οι μεσογειακές χώρες. Ο κύριος Νόιζερ αναφέρθηκε στις κοινοβουλευτικές διασκέψεις. Εγώ έχω να σας πω ότι το Κρατικό Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στις εργασίες αυτές και γίνονται ανταλλαγές με τις αρμόδιες αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα υπάρχουν όλο και περισσότερες. Τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα καλά τα τελευταία στοιχεία της ερώτησής σας για την πρόοδο στα Δυτικά Βαλκάνια. Πάντως, αν θέλουμε μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλουμε πραγματικά να αποτελούμε παράγοντα υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας παγκοσμίω, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε τι γίνεται στη δικιά μας περιοχή. Η ειρήνη και σταθερότητα διότι ό,τι έχουν πετύχει η Κροατία, η Σλοβανία αποτελούν παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες, για τις χώρες αυτές των Δυτικών Βαλκανίων και τους δείχνει ότι και εκείνες μπορούν να φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εγωιστές, μπορούμε να μοιραζόμαστε την πραγματογνωμοσύνη μας, τις εμπειρίες μας και εμείς ασπαστήκαμε πλήρως τι αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχεί. Βλέπουμε πόσο πολλοί τουρίστες έρχονται στην Αδριατική θάλασσα, αλλά δεν είναι κροατική η Αδριατική θάλασσα, είναι ευρωπαϊκή. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ελπίζω να μπορούμε να βασιστούμε και στη δικιά σας στήριξη για να ενταχθούμε στο χώρο του Σέγγεν. Νομίζω ότι αυτό απαντάει στην ε, ερώτησή σας. Έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως, είπε ότι καλύπτει και το 8 κριτήρια η Κροατία για να ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν. Είμαστε λοιπόν περήφανοι για τη στάση της κροατικής αστυνομίας στο θέμα της προστασίας των συνόρων μας απέναντι στην οργανωμένη εγκληματικότητα και αυτό ίσως να απαντάει και στην ερώτησή σας για τη μετανάστευση. Για να προστατέψει λοιπόν η αστυνομία μας τα παράνομα μεταναστευτικά ρεύματα. Μία προτεραιότητά μας λοιπόν είναι η Ευρώπη η οποία προστατεύει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύεται από την παράνομη μετανάστευση και την τρομοκρατία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, να σας αποχαιρετήσω και στα γερμανικά γιατί ήταν πριν από λίγες μέρες στην πρεσβεία μας στο Βερολίνο. Ε, νομίζω ε, μπορώ να πω από καρδιάς εκ μέρους όλων των ευρωβουλευτών εδώ. Καλή τύχη για το εξάμεινό σας. Ακούσατε όλα τα μέλη να παίρνουν εδώ το λόγο για να σας πούν ότι σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς στα πλαίσια της παγκόσμιας κρίσης, των παγκόσμιων κρίσεων έχουμε πολλά να κάνουμε. Ελπίζουμε λοιπόν στη Σύνοδο στα Βαλκάνια αρχές Μαΐου να ε, έχουμε ακόμη περισσότερο καλό ρυθμό για την ε, υλοποίηση της πολιτικής μας και την συνέχισή της και ως γειτονική χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια μπορείτε να προσφέρετε τις ειδικές σας τεχνικές γνώσεις και ε, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και καλή τύχη για την κρατική προεδρία.